Um, it is now 10 o'clock. Uh, we should start this hearing. Είναι 10 η ώρα να αρχίσουμε. Γιατί έχουμε πολλά. Παρακαλώ, καθίστε όλοι. Σας παρακαλώ, καθίστε πρέπει να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε, είναι κοινή ακρόαση μεταξύ της ΣΥΝΤΑ και της Επιτροπής Γυναικών και με χαρά συμπροεδρεύω με την αντιπρόεδρο της ΣΥΝΤΑ, την κυρία Σαΐφη, εδώ αριστερά μου. Η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μας ήταν πάντα έξοχη και ελπίζω η εργασία για το σημαντικό αυτό θέμα που είναι η ισότητα των φύλων ε, να προωθηθεί. Η προώθηση τη ισότητα των φύλων ήταν πάντα βασική προτεραιότητα τη Ένωση από την αρχή. Όμω, σε ορισμένου τομεί πολιτική, ιδιαίτερα στην εμπορική πολιτική, δεν έχουμε πλήρω ε, επιτύχει αυτό το στόχο. Οι συμφωνίε εμπορίου και επενδύσεων έχουν διαφορετικά αποτελέσματα στι άντρε και τι γυναίκε και διάφορε μελέτε έχουν σαφώ αποδείξει ότι το εμπόριο δεν είναι ουδέτερο από πλευρά φύλου. Πρέπει λοιπόν να το αναλύσουμε από Πλευρά φίλου. Να δώσω το λόγο στην συμπρόεδρό μου, την κυρία Ζέιφη. Ευχαριστώ, κυρία Αντιπρόεδρε. Καταρχάς, ε, να καλωσορίσω τις ε, εμπειρογνώμονες που είναι ε, σε αυτήν την εκδήλωση σήμερα μαζί μας και χαίρομαι που συμπροεδρεύω μαζί με την κυρία Χάλιμπο που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών. Είμαι πεπισμένη ότι η κοινή μας εργασία για το θέμα αυτό θα ε, φέρει καρπούς. Ε, σήμερα θέτουμε το θέμα της ισότητας ανδρών γυναικών στις ε, εμπορικές συμφωνίες. Πώς μπορεί να συμπεριληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης. Είναι πολύ επίκαιρο θέμα, διότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων για τον εξυγχρονισμό της εμπορικής συμφωνίας με τη Χιλή. Χαίρομαι πολύ για αυτήν την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι σήμερα παρούσα να μας δώσει περισσότερες προφορίες για το θέμα αυτό. Γενικότερα και λόγω των επιπτώσεων του εμπορίου επί της οικονομίας γενικότερα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα θέματα φύλου και ισότητας φύλου στην ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Έχουμε ε, και επίσης τι μελέτες αντικτύπου στις διαπραγματεύσεις κάθε εμπορική συμφωνία θα έπρεπε να λαμβάνει <clears throat> υπόψη το θέμα του φύλου. Η ισότητα ανδρών γυναικών είναι μια ευκαιρία για να υπάρξει καλύτερη κατανομή των ωφελών από μια συμφωνία. Να ωφελούνται όλοι. Θα πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν αυτό το θέμα και είμαι πεπισμένη ότι οι συζητήσεις που θα έχουμε με τους ε, εμπειρογνώμενε θα είναι επικοδομητικέ. Να δώσω το λόγο λοιπόν στην πρώτη ομιλήτριά μα, την κυρία Μάρτσια Φοντάνα που είναι οικονομολόγος που ασχολείται ιδιαίτερα με τα θέματα ισότητας ε, ανδρών γυναικών στο διεθνές εμπόριο ιδιαίτερα και την οικονομία γενικότερα. Κυρία Φοντάνα, έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Γενικές παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα για τη σχέση μεταξύ φύλου και εμπορίου με βάση τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής και μετά θα πω ότι πρέπει να υπερβούμε την εξέταση απλώς της ε, φιλελευθεροποίησης της αγορα... Ε, των... Ε, του εμπορίου αγαθών. Πρέπει να δούμε τι ρόλο παίζει και η φιλελευθεροποίηση των κανονισμών, των υπηρεσιών και των προδιαγραφών. Γιατί είναι σημαντικά στοιχεία των συμφωνιών που έχουμε τώρα, των ισχυουσών. Και κατόπιν να κάνουμε και μερικέ προτάσει γιατί τι μπορεί να κάνει η Ένωση για να διασφαλίσει ότι οι εμπορικέ συμφωνίε ακριβώ περιλαμβάνουν στόχου ισότητα φύλων. Πρώτον, να διευκρινίσω. Ορισμένοι μπορεί ακόμη να πιστεύουν ότι δεν παίζει ρόλο το θέμα του φύλου στην εμπορική πολιτική. Είναι σαφέ όμω ότι ισχύει το αντίθετο, το αντίθετο. Γιατί το εμπόριο λειτουργεί εντό οικονομιών. Οι οποίε οικονομίε ε, κάνουν διακρίσει κατά των γυναικών. Οι γυναίκες είναι σε άλλε απασχολήσει από τους άντρε, κυρίως σε επισφαλείς μορφέ εργασίας, αντιμετωπίζουν ε, ε, περισσότερες ευθύνε ε, για τι τις εργασίε και δεν είναι μόνο χρονικέ αυτές οι απαιτήσει, αλλά έχουν και περιορισμό στην πρόσβαση σε πηγές παραγωγής όπως είναι η γη και η πίστη. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την κατάσταση. Και έχουμε πολλά στατιστικά στοιχεία που στηρίζουν ε, την προσπάθειά μας αυτή. Αυτό έχει να κάνει ε, και ισχύει για όλες τις χώρες, είτε υψηλών είτε χαμηλών εισοδημάτων και έχει δύο επιπτώσεις για τον τρόπο με τον οποίο ε, το φύλλο και το εμπόριο αλληλεπιδρούν. Η πρώτη επίπτωση είναι ότι υπάρχουσα ανισότητα, υπάρχουσα, υπάρχουσα ανισότητα παίζει ρόλο στην ανταγωνιστικότητα και τελικά και οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις παίζουν ρόλο. Δηλαδή ε, τελικά η ανισότητα του φύλου έχει κακό αποτέλεσμα και στην ε, ε, αποδοτικότητα του εμπορίου. Για παράδειγμα στην Ασία έχουμε διαπιστώσει ότι παίζει ρόλο αυτό διότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις γυναίκες που πληρώνονται χαμηλά για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα των χωρών. Αυτό όμως έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Γιατί μακροπρόθεσμα αποθαρρύνει την ε, τεχνική καινοτομία και την ανάπτυξη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Ναι, ναι, θα μιλήσω λίγο πιο αργά. Σε άλλες περιπτώσεις, η ανισότητα φύλου, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν πρόσβαση γυναίκες στην ε, γη και τις αγορές σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στις ε, προκλήσεις ε, προσφοράς η οικονομία και η γεωργία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται αυτή η ανισότητα. Για παράδειγμα, η απασχόληση. Εδώ έχουμε τα περισσότερα στοιχεία και αυτό συζητάμε. Αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η ανισότητα και μέσω τη κατανάλωση και τη παροχή δημοσίων υπηρεσιών. Διότι οι δημόσιες υπηρεσίες ε, παρέχονται διαφορετικά φύλλο και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Σε πολλές χώρες ορισμένες υπηρεσίες παραδοσιακά ε, ήταν δημόσιες. Το ρόλο και περισσότερο υπόκειται σε ανταγωνισμό από ξένες εταιρείε. Ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν για την απασχόληση. Βεβαίω υπάρχουν διαφορές αναφύλων, διότι στου εμπορεύσιμου και, και μη εμπορεύσιμου ε, τομείς είναι διαφορετική η κατανομή της απασχόλησης. Άρα δεν μπορεί να υποκαταστήσει ε, η απασχόληση ε, μέσω ενός φύλου την απασχόληση του άλλου. Ξέρουμε ότι στον αναπτυσσόμενο κόσμο οι γυναίκες έχουν ε, επωφεληθεί από θέσει εργασία που σχετίζονται με το εμπόριο αλλά μόνο σε χώρες όπου αναπτύχθηκε ε, η ελαφρά βιομηχανία, όχι σε χώρες που έχουν άλλες εξαγωγικές δομές. Αλλά ακόμη και στον κατασκευαστικό τομέα, οι γυναίκες έχουν περιοριστεί σε χαρακτηριστικά ε, γυναικείες δουλειές που είναι συνήθως επισφαλείς. Επίσης ε, έχει επιπτώσεις αυτό και στον τρόπο κατανάλωσης. Αυτό τι σημαίνει. Οι γυναίκες έχουν την κύρια ευθύνη για την αγορά, και την προετοιμασία του φαγητού για τις οικογένειές τους. Ε, μία από τις επιπτώσεις του, της ναύτα, για παράδειγμα, ήταν, ήταν ότι αυξήθηκε η τιμή των τοπικά παραγωμένων τροφίμων, ενώ μειώθηκε η τιμή ε, χαμηλής ποιότητας τροφίμων που εισάγονται από τις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι ε, επιδεινώθηκε η ποιότητα της διατροφής πολλών παιδιών στο Μεξικό. Επίσης, η αλλαγή των δημοσίων δαπανών λόγω του εμπορίου παίζει ρόλο επίσης και έχει επιπτώσεις ε, διαφορετικές στα δύο φύλλα. Αυτό ισχύει και με τις αισχύουσε εμπορικέ ε, συμφωνίε όπως την ε, ΣΕΤΑ. Δεν υπάρχει ισότητα πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και στην ποιότητα της παροχής. Σε χώρες υψηλού και μέσου εισοδήματος η απελευθέρωση, για παράδειγμα, τη ε, της ιατρικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους ε, θα θίξει περισσότερο τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο, αλλά είναι ε, φτωχότερες από τους άντρες και παίζουν περισσότερο ρόλο στη φροντίδα που παρέχεται για τους ηλικιωμένους στην οικογένεια. Σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, η ιδιωτικοποίηση της ίδρυυσης επίσης μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Γιατί οι γυναίκες και τα κορίτσια όπως ξέρουμε που συνήθως πηγαίνουν και ε, να πάρουν νερό εκεί που δεν υπάρχει ε, πρόσβαση σε πόσιμο νερό μέσω δικτύου. Βεβαίως ε, μπορεί να υπάρξουν περισσότερες ε, δυνατότητες ε, απασχόλησης των γυναικών στις κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί εδώ κυ κυρίως εργάζονται γυναίκες. Αλλά αν δεν υπάρχει επαρκής οικονομική στήριξη από τις κυβερνήσεις, η φιλελευθερωποίηση και η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών μπορεί να σημαίνει ότι τελικά οι δημόσιες παροχές μπορεί να αντικατασταθούν από ιδιωτικού τύπου υπηρεσίες που θα είναι προσβάσιμες μόνο σε όσους μπορούν να τις πληρώσουν. Οπότε κλείνοντας αυτό το σημείο, όλα αυτά τα αποτελέσματα με όλους αυτούς τους τρόπους μπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά. Το εμπόριο δεν είναι περσέ θετικό ή αρνητικό, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ε, σχεδιάζονται οι εμπορικές πολιτικές. Τώρα οι ενωσιακές ε, εμπορικές πρακτικές και συμφωνίες. Η Ένωση έχει υπογράψει εμπορικές συμφωνίες με χώρες και του Βορρά και του Νότου. Το ΣΕΤΑ, με το, ή ΣΕΤΑ με τον Καναδά για παράδειγμα. Ενώ οι, οι, οι συμφωνίες ΕΠΑ, οι συμφωνίες συνεργασίας και εταιρικής σχέσης με χώρες του Νότου ε, είναι παράδειγμα συμφωνιών λοιπόν με τις χώρες ακριβώς του Νότου. Σε ένα πρόσφατο κείμενο, ε, μια πρόσφατη εργασία που σας απέστειλα τον προηγούμενο Νοέμβριο εδώ στην Επιτροπή σας, θα παρουσιάζω αυτά. Το σημαντικό είναι να δούμε τι ρόλο παίζουν αυτές οι εμπορικές συμφωνίες για την ισότητα των φύλων, όχι μόνο στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά και σε τρίτες χώρες, με τις οποίες έχει εμπορικές σχέσεις η Ένωση, ιδιαίτερα στον αντισώμενο κόσμο. Και πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξουν ε, εμπορικοί κανόνες που να σέβονται τα ε, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των γυναικών. Η ΔΕΟΔΟΣ, η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει να προσεχθεί περισσότερο η ισότητα των φύλων σε κάθε φάση της ε, διαμόρφωσης τη εμπορικής πολιτικής. Όταν συλλέγονται στοιχεία για να βασιστούν οι αποφάσεις για τις εμπορικές συμφωνίες, όταν σχεδιάζεται η πολιτική, όταν γίνονται οι διαπραγματεύσεις και για να βοηθάμε την εφαρμογή επιτόπου για να εφαρμοστεί σωστά. Πρέπει να βελτιωθεί συγκεκριμένα η ποιότητα των μελετών αντικτύπου που γίνονται. Και στη μελέτη μου αναφέρομαι ιδιαίτερα στη μελέτη αντικτύπου της ΣΕΤΑ. Θα ήταν σημαντικό να έχουμε περισσότερα στοιχεία για τι επιπτώσεις έχουν στην ισότητα φύλου οι αλλαγές στις υπηρεσίες, προδιαγραφές και τους κανονισμούς. Και θα πρέπει η ανάλυση φύλου να συμπεριλαμβάνεται στην παρακολούθηση της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών μετά την υπογραφή τους. Στη φάση των διαπραγματεύσεων η Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις για φιλελευθερωποίηση να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των γυναικών. Δεν υπάρχει μία ε, εμπορική πολιτική που να είναι κατάλληλη για όλες τις περιστάσεις. Πρέπει να σχεδιάζεται η εμπορική πολιτική ούτω ώστε να διασφαλίσει ότι τα οικονομικά και, δικαιώμα... και κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών και άλλων ευαλότων ομάδων λαμβάνονται υπόψη. Παράδειγμα, οι διαπραγματευτέ θα πρέπει να έχουν ένα κατάλογο των τομέων ε, όπου παίζει μεγάλο ρόλο το θέμα του φύλου, ούτω ώστε, για παράδειγμα, να υπάρξουν εξαιρέσει από τη ελευθεροποίηση ή, ή μεταβατικέ περίοδοι και οι νέε συμφωνίε ε, εμπορίου και επενδύσεων πρέπει να εξετάζονται και από πλευρά των επιπτώσεων που έχουν στις προδιαγραφέ και του κανονισμού. Υπάρχουν πολλά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό οποιασδήποτε ε, προβλέψεις, οποιαδήποτε μέτρα να μην υπονομεύουν ε, τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να προωθήσουν την ισότητα φύλου. Πρέπει να υπάρξουν επίσης αποτελεσματικά μέτρα από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για να αποζημιωθούν οι ομάδες εργαζομένων και καταναλωτών που θα υποστούν βλάβη από κάποιες συμφωνίε Πολύ συχνά προβλέπονται στα λόγια, στα χαρτιά αυτά τα μέτρα, αλλά η εφαρμογή τους μέχρι στιγμής υπήρξε ιδιαίτερα ανεπαρκής. Στο επίπεδο εφαρμογής μετά των συμφωνιών ιδιαίτερα συμφωνών εμπορίου με αναπτυσσόμενε χώρε η Ένωση θα μπορούσε να αξιοποιήσει το πλαίσιο της ε, πολυμερούς ε, βοήθεια για την ανάπτυξη για να βοηθήσει τι κυβερνήσει των χωρών αυτών για να εφαρμόσουν του στόχου ισότητα των φύλων στα πλαίσια της ε, εμπορική στρατηγική του. Να σταματήσω εδώ και βεβαίως θα τα πούμε μετά στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Φοντάνα για αυτήν την πλήρη παρουσίαση. Νομίζω ότι μας βοηθά πάρα πολύ σε όλα αυτά που πρέπει να μάθει και τώρα. Έχει η κυρία Μαρία Μαγούλιαμς, η οποία είναι ανώτερη υπάλληλο στο κέντρο του Νότου, South Center της Γενέβης και ασχολείται με θέματα όπως η χρηματοοικονομική κρίση, η αλλαγή του κλίματος, η χρηματοδότηση της σχετικής πολιτικής και τα θέματα ανάπτυξης επίσης έχει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά το κρατικό χρέος και το διεθνές εμπορίο και το λόγο για 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ και καλημέρα εις όλους και ευχαριστώ και τις δύο επιτροπές σας διότι με καλέσατε να συμμετάσχω σε αυτή την σημαντική εκδήλωση περιμένω πώς και πώς να τα συζητήσουμε ακριβώς όπως και η κυρία Φοντάνα που είπε τόσα και ουσιαστικά για τα δύο φύλλα, την ισότητα των δύο φύλων και το εμπόριο. Εγώ να σας πω τι γίνεται όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά πρώτα θέλω να αρχίσω με κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται για ένα έγγραφο τη Διεθνού Τράπεζα, του ε, Διεθνού ε, Νομισματικού Ταμείου, του, του Μάρτιο ε, συνετάχθη και λένε αυτοί οι οργανισμοί ότι η εμπορία αφήνει πίσω πάρα πολλού και πάρα πολλέ οικονομίε, κυρίω στι προχωρημένε, προοδευμένε κοινωνίε, οπότε υπάρχει οικονομικό μειονέκτημα ε, και πολλές φορές ε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκληρά και αυτές οι συνέπειες ε, κρατούν πολύ και μετά σε αυτό το έργο αναγνωρίζουν το τι γίνεται όσον αφορά το, το εσωτερικό εμπόριο και ότι θα, θα μπορούσε η διεθνή συνεργασία να βοηθήσει όμως ούτω ώστε με κάποιες διατάξεις δικαίου προαιρετικές και κάποιες άλλες συμφωνίες, να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ιδιορυθμίες, να υπάρξει διάλογος και συνεργασία στην μακροοικονομική πολιτική, ούτω ώστε να βοηθηθούν οι εσωτερικέ πολιτικές. Αυτά λοιπόν ε, είναι αυτά που λένε οι ακτιβιστές εδώ και 20 και πάνω χρόνια. Αλλά δεν τους ακούνε πολλοί αυτοί οι οποίοι χαράζουν τις ε, πολιτικές. Και επομένως βλέπουμε το πόσο σκληρό είναι το εμπόριο και στη ΣΥΠΑ και στον Εμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε δει πολλές εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου. Όντως ήρθε η ώρα ούτω ώστε να καλύψει το θέμα της όντας των φίλων και το εμπόριο. Έχουμε και αυτή τη συμφωνία με την ε, Χιλή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε και αυτά θα πρέπει εκεί να ληφθούν υπόψη. Τώρα, για να μην το ξεχάσω, να σας πω για τέσσερις τομείς που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως είπε η κυρία Φοντάνα. Βεβαίω ε, το θέμα του, της ε, βοήθειας μέσω του εμπορίου 200 δις δολάρια και 3% όμως ε, αφορούσαν την ισότητα. 1,3 δις δαπανήθηκαν το 2011 Οπότε αυτό το aid for trade θα πρέπει να επανασχεδιαστεί και να προσανατολιστεί και προς την ισότητα των φύλων. Επίσης, στις νέες κατευθύνσεις ε, που αφορά την ισότητα των φύλων και την έρευνα είναι αυτό που μας είπε και η κυρία Φοντάνα. Νέους τομείς όπου θα πρέπει να υπάρξει ε, παρέμβαση και ελπίζω και εσείς θα τα λάβετε υπόψη όταν έχουμε αυτές τις συμφωνίες διευκόλυνσης της εμπορικές που από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη σχέση με τον ΠΟΕ, τι γίνεται με τις γυναίκες και τις μη μη έψιλον. Ε. Και υπάρχει ένας μύθος ότι κάπως οι γυναίκες καλύπτονται από την αξιακή αλυσίδα. Μύθος. Επίσης, το πόσο όλοι θέλουμε να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και εκτός από την ισότητα των φύλων, εδώ είναι και θέμα εμπορίου. Αυτή η στόχη, επομένω, που έχει τάξει την εμπορική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το εμπόριο για όλους. Άρα θα πρέπει έτσι να συνδέσουμε εμπόριο και ισότητα των φίλων. Και τώρα το τελευταίο που θέλω να σας επισημάνω είναι κάτι το οποίο προκύπτει στη συζήτησή μας πέραν της χρηματοοικονομικής κρίσης και της ε, ανάκαμψης είναι η περιβαλλοντική κρίση. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς επηρεάζονται οι γυναίκες από τις αλληλένδετες επιμέρους διαφορετικές πολιτικές. Τώρα για να σας πω αυτά τα οποία έχω προετοιμάσει ως παρουσίαση. Ξέρω ότι έχω μόνο 7 λεπτά και λέμε για το πώς οι εμπορικές πολιτικές επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα είπε η κυρία Φοντάνα, είναι πολύ σημαντικά για την προβληματική μας. Οπότε για να μην σας κουράσω, αλλά είχα να πω ότι βεβαίω και οι γυναίκες αντισώμενες χώρε καλύπτονται από τις ε, εμπορικές ε, δραστηριότητε, είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο τους και για τις εξαγωγές, αλλά έχουμε θέματα ε, ισότητα των φίλων, τη χειραφέτηση των γυναικών, όλα αυτά είναι αλληλένδετα όσον αφορά την επέκταση, τη διεύρυνση του εμπορίου και την εντατικοποίηση του εμπορίου. Γιατί υπάρχει εδώ και το θέμα του μισθολογικού χάσματος, η επίδραση στις μικροεπιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις, γιατί μιλάμε για 40-50% αυτών των επιχειρήσεων που καλύπτονται προβλήματα, προκλήσεις για την καθημερινή ζωή των γυναικών. Τώρα όσον αφορά τις ε, πολιτικές εμπορίου των, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και επίσης και το GSP Plus. Έχουμε διάφορα είδη συμφωνιών. Έχουμε την αρχή everything but arms, όλα να είναι αντικείμενο εμπορίου αλλά όχι όπλα για τις αντισώμενες χώρες και η σχέση ε, αυτής της αρχής με τον ΟΕ. Οπότε έτσι έχουμε την κοινή ε, γεωργική πολιτική, έχουμε τις επιδοτήσεις, αλλά επίσης έχουμε τα ελάχιστα εργασιακά πρότυπα. Αχ, δεν μπορώ τώρα λήψη χρόνου να μπω στις λεπτομέρειες, να σου πω, πω τι επιπτώσεις υπάρχουν για την ισότητα των φύλων από αυτά. Πάντως θέλω τώρα να επισημάνω τις εξής τρεις πτυχές του θέματος. Ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ε, Ένωσης έχουν σχέση με τις ε, επιπτώσεις για τις ΜΜΕ. Επίσης ε, η κρατική πολιτική που αφορά τις υπηρεσίες και την απελευθέρωση σχετικής πολιτικής, επίσης όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και έχουμε τις τελευταίες διατάξεις όσον αφορά την επίλυση εμπορικών διαφορών στα πλαίσια και των εμπορικών συνθήκων. Και μιλάμε για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τι κάνουν εκεί οι γυναίκες επιχειρηματίες. Ε, και θεωρούμε ότι εκεί με μαγικό τρόπο ρυθμίζονται όλα, αλλά φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και συχνά αυτές οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θίγονται από τις εμπορικές συμφωνίες. Απαγορεύεται από τις εμπορικές συμφωνίες να υπάρξει κυβερνητική στήριξη σε αυτές τις επιχειρήσεις των γυναικών. Και αυτό γιατί θεωρείται ότι μπορεί να επισύρει αγωγές και να αντιβαίνει στις εμπορικές συμφωνίες. Μα είπε επίση και γι' αυτό η, η Δ. Φοντάνα. Επίση, να δούμε τι γίνεται στι δημόσιε συμβάσει, είναι ένας από τους τρόπους που οι αναπτυσσόμενες χώρες προσπαθούν να αποκαταστήσουν κάποια έλλειψη ισορροπιών, κάποιου είδου ιστορικές ε, διακρίσεις κατά των Ιθαγενών στην Νότια Αφρική και κατά των γυναικών. Οπότε αυτές οι συμβάσεις τώρα ε, είναι ένα... υπάρχει κάποιο φρένο τέλος πάντων τι μπορεί να κάνει το ε, το κράτος για να βοηθήσει σε περισσότερη ισότητα. Γνωρίζουμε επίσης ότι επίσης, ε, επίσης έχουμε και ε, τους ανάπηρους οι οποίοι και αυτοί θα έπρεπε να ευνοούνται από το κράτος και σε περίπτωση που έχουν κάποιες επιχειρήσεις. Μια που όλα αυτά επομένως αλληλοσυνδέονται, συνδέονται τι γίνεται, ότι κάποιες γυναίκες μπορεί να είναι φτωχές, κάποιες άλλες μπορεί να είναι άπειρες και θα πρέπει να αναλυθεί το πώς επηρεάζονται αυτές οι γυναίκες. Και έχουμε την Συμφωνία Συναλλαγής Υπηρεσιών, την ΤΙΣΑ, που αφορά τις αμοιβέ των γυναικών, το τι γίνεται και με απορρίθμιση στις υπηρεσίες ε, έχουν καταλήξει σε φτώχεια οι γυναίκες και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα για το πώς η αχαλήνωτη απελευθέρωση έθιξε τις γυναίκες και γνωρίζουμε ότι στις, στην Ευρώπη ε, οι κρατικές υπηρεσίες έχουν αναλυφθεί από τις τοπικές αρχές οπότε υπάρχει ακόμα λιγότερο έλεγχο του τι γίνεται σε αναπτυσσόμενες χώρες. εν κατακλείδη να σας πω τι γίνεται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Συμφωνώ με την Δ. Φοντάνα ότι αυτοί που χράσουν την πολιτική και αλλά και την εμπορική πολιτική θα πρέπει να κάνουν κάποιο είδου παρεμβάσεις ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη ο ρόλος της γυναίκας για την οικονομία σε σχέση με τον άνδρα και στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να γίνει μια τέτοια επανέμβαση που να διευκολύνει την οικονομική κινητικότητα σε περισσότερου τομεί και σε περισσότερα επαγγέλματα και να έχουν περισσότερε επιλογέ οι γυναίκε. Οπότε το θέμα είναι ποιο είναι ο ρόλο πώ μπορεί να συμβάλλει στην ισότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι εμπορικέ συμφωνίε, ιδίω όσον αφορά τι χώρε ΑΚΕ. Και εδώ υπάρχουν ε, προκλήσει αλλά και ευκαιρίε, μα τα είπε η δόκτωρ Φοντάνα τι γίνεται με την κατανάλωση, με την απασχόληση, τι γίνεται με τις υπηρεσίες, αλλά επίσης υπάρχουν και ευκαιρίες από την εμπορική συμφωνία για να υπάρξει ανάπτυξη και όχι μόνο να εκμεταλλεύει κανεί τους ε, πόρους και να διονύζει τη φτώχεια. Οπότε έτσι θα πρέπει να δούμε το θέμα. Να γίνει αξιολόγηση του πώς όλα αυτά θα υλοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ σκληρή με τις αφρικανικές χώρες για να ε, υπογράψουν τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης της ΕΠΑ. Ε, μπήκε η προθεσμία του Οκτωβρίου, θα είχαν τα προνομιά τους να δεν ε, υπέγραφαν της ΕΠΑ, οπότε τώρα αρχίζει το θέμα του όταν τεθεί σε εφαρμογή η ΕΠΑ τι θα κάνει ο κόσμος στις χώρες εκείνες, άντρες και γυναίκες. Οπότε θα πρέπει να δει κανεί το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τη ΣΕΠΑ. Οι οικονομολόγοι και οι τράπεζες λένε τι στοιχεία έχετε. Με τη ΣΕΠΑ τώρα μπορούμε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και επίσης κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για να δούμε προς τα πού θα πάμε με τις ΕΠΑ. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, κυρία Williams. Και τώρα η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Χέα Μάιερς. Από ε, το White Plus. Ε, για θέματα ισότητα ανδρών και γυναικών στην οικονομία και στην πολιτική ανάπτυξη. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τις Επιτροπές ΣΥΝΤΑ και ΕΦΕΜ που με προσκάλεσαν, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι οργανώνουν αυτή τη σημαντική ακρόαση ε, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και μια ευκαιρία να το συζητήσουμε τώρα τη στιγμή που γίνονται τόσες ε, διαπραγματεύσεις ε, σχετικά με το εμπόριο. Σας εκπροσωπώ εδώ πέρα το White Plus και ορισμένα από τα πράγματα τα οποία θα αναφέρω σήμερα έχουν ήδη συζητηθεί από την κυρία Φοντάνα και Williams όμως θα ήθελα εδώ να σας παρουσιάσω το δίκτυό μας το οποίο εκπροσωπεί κοινωνίες των πολιτών σε 10 χώρες στην Ευρώπη. Ε, και αθώς επίσης και έχουμε ε, εταίρους ε, στον Νότο. Ασχολούμαστε εδώ και πάνω από 20 χρόνια με τις εμπορικές συμφωνίες από τις άποψεις των, από πλευράς σε ζητήματα φύλου. Η εμπειρία μας έχει ότι παρακολουθώντας τις εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα τελευταία ε, χρόνια, η ε, ευρωπαϊκή πολιτική εμπορία είναι ε, τυφλή από άποψη φύλου και αυτό το σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνει πιο περιεκτική όσον αφορά τα ζητήματα φύλου, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι είναι και ιδιαίτερα νεοφιλελεύθερη ε, μια, ε, ακολουθεί πολιτική που προωθεί την κατάργηση των διεθνικών ε, δασμών, την απορρίθμιση των επενδύσεων και των υπηρεσιών, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επενδυτών και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και προστατευτικές πολιτικές ιδιαίτερως απέναντι στους Ευρωπαίους παραγωγούς αλλά και σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ε, το έχουμε δει αυτό και σε άλλες ε, χώρες ε, της Δύσης όπου προωθείται κάτι τέτοιο και βλάπτει ιδιαίτερο στην βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα των γυναικών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διαφορετική πολιτική κατά τη γνώμη μας. Έχουν γίνει πολλές έρευνες όμως ε, υπάρχει και ε, εμπειρική έρευνα σχετικά με συμφωνίες ελεύθερου, ελεύθερων συναλλαγών και ε, στο πλαίσιο του ΟΗΕ ανησυχούν για τις υπάρχουσες πολιτικές. Βλέπουμε λοιπόν περιπτώσεις φτωχών γυναικών ή θα γινών γυναικών, γυναικών με μεταναστευτικό υπόβεθρο που επηρεάζονται ιδιαίτερως από τις συγκεκριμένες πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να προωθήσει την ισότητα των φύλων το οποίο αποτελεί ε, αναπόσπαστο κομμάτι της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και στις αναπτυξιακές πολιτικές υπάρχει ε, πολύ έργο σχετικά με την ισότητα των φύλων πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε. Ήδη το 2006 στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου υιοθετήθηκε μια απόφαση σχετικά με τις γυναίκες διεθνές, με το διεθνές εμπόριο. Πολλές από τις προτάσεις που έγιναν πριν από αρκετά χρόνια ισχύουν ακόμα το 2017 ε, και εμείς ε, το ε, υποστηρίζουμε όλο αυτό. Και τώρα θα επαναλάβω κάποια από τα πράγματα τα οποία έχουν ήδη υποθεί από την κυρία Φοντάνα και Βίλιαμ σχετικά με το εμπόριο. υπάρχει ή ε, ε, γενικότερα ε, το, στο, στο εμπόριο βλέπουμε ότι πλήττονται ιδιαίτερως οι γυναίκες όσον αφορά την απελευθέρωση του εμπορίου. Θεωρούμε επίσης ότι αυτή η ανάπτυξη με βάση τις ε, εξαγωγές έχει επηρεάσει ιδιαίτερα στις γυναίκες οι οποίες πληρώνονται λιγότερο κάτω από τα αξιοπρεπή επίπεδα ε, κάτω από επίπεδα τα οποία μπορούν να τους χαρίσουν ένα ε, βιώσιμο τρόπο ζωής επανερχόμενοι στα όσα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τη Συμφωνία εμπορίου έχει κάνει ε, προσφάτως όσον αφορά το φύλλο. Έχουμε γεγονότα τα οποία επικεντρώνονται στη χειραφέτηση των γυναικών σχετικά με το εμπόριο. Στις 20 Ιουνίου θα έχουμε μια συνάντηση πάνω σε αυτό και έχουμε επικεντρωθεί ιδιαιτέρως ε, στην επιχειρηματικότητα των ε, γυναικών ε, που θα πρέπει να προωθηθεί στο εμπόριο για να προωθήσουμε με αυτόν τον τρόπο την ισότητα των φίλων στο εμπόριο. Χαιρετίζουμε επίσης οποιαδήποτε πρωτοβουλία η οποία θα προωθήσει την ισότητα των φίλων, όμως θεωρούμε ότι, θα πρέπει να ότι επικεντρωνόμαστε μονάχα στην επιχειρηματικότητα των γυναικών που όμω αποτελούν μονάχα ένα μικρό ποσοστό των εργαζομένων γυναικών οι περισσότερες εργάζονται στον ανεπίσημο τομέα αλλά και στη γεωργία κάνοντας άμυστη εργασία, ε, φροντίζοντας τις οικογένειες ε, για ε, παράδειγμα. Επίσης ασχολούνται εποχικά και οι γυναίκες αυτές είναι αόρατες στις εμπορικέ συμφωνίες παρόλο όμως που παράγουν ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομικής παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, διευρύνουμε ε, την σκοπιά μας πάνω σε αυτό και να μην επικεντρωνόμαστε μονάχα στις γυναίκες επιχειρηματίες. Με βάση λοιπόν όλο αυτό το όραμα θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μονάχα στην προώθηση ε, της ε, γυναικείας επιχειρηματικότητας ε, στο επικεντρώτο και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, όμως θα πρέπει να προσθέσουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίων και τι είδους θέσεις εργασίας και ευκαιρίες δημιουργούνται, διότι αυτές θα δημιουργήσουν σε αξιοπρεπή εργασία και ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Ε, ε, έχουμε, δεν θα πρέπει να υπάρχει σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, θα πρέπει να υπάρχουν σωστές συνθήκες εργασίας. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προσταθούν όταν, εργαζόμαστε, όταν ασχολούμαστε με την επιρροή των συμφωνιών εμπορίου που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να ε, προσθέσουμε κεφάλαια ε, βιωσιμότητας, να προσθέσουμε τα πρότυπα του Άιλο όσον αφορά τις γυναίκες όπως ήταν η ε, συμφωνία, ε, η σύμβαση 189 και 156 ε, σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες, όπως επίσης έχουμε και την σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάρτηση όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών Όλα αυτά τα εργαλεία λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα ε, κεφάλαια ε, βιωσιμότητας ε, και θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στα βασικά κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά θα αποτελέσουν ένα σημαντικό κομμάτι των κεφαλαίων για το εμπόριο όπως επίσης και στην περίπτωση ε, της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ε, που διαπραγματευόμαστε με τη Χιλή. ιδιαίτερο επειδή θα πρέπει να διασφαλίσουμε αξιοπρεπέ συνθήκε εργασίας ε, για τις ε, γυναίκες, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Οι προηγούμενοι ομιλητέ είπαν κάποια πράγματα σχετικά με τις ε, συνέπειες της Ευρωπαϊκή Πολιτική εμπορίου ε, που ε, έχει οδηγήσει σε απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου καταργώντας και μειώνοντα τους δασμούς και προωθώντας την απελευθέρωση των αγορών υπηρεσιών και επενδύσεων μεταξύ αυτών και των δημοσίων συμβάσεων ε, συμφωνούμε ότι οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα από την απελευθέρωση των ε, υπηρεσιών και δημοσίων συμβάσεων και θα θέλουμε να προσθέσουμε ότι παγκοσμίω οι γυναίκες περνούν δυόμιση φορές περισσότερο ε, χρόνο εργαζόμενες άμυστα για να φροντίζουν τις οικογένειές τους σε σχέση με τους άνδρες κάτι το οποίο έχει ερευνηθεί ευρέως ε, η δουλειά αυτή γίνεται κυρίως από τις ε, γυναίκες ε, και δεν συμπεριλαμβάνεται αυτή η συνεισφορά των γυναικών στις οικονομίες, όμως πρόκειται για έναν μεγάλο οικονομικό τομέα και κατά τη γνώμη μας το άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών και δημοσίων συμβάσεων ε, εμποδίζουν την πρόσβαση σε ε, βασικές ε, κοινωνικές παροχές με αποτέλεσμα να, κάνουν, να επιβαρύνονται ιδιαίτερως οι γυναίκες. Επίσης, σε σχέση με όλα αυτά, όταν έχουμε απελευθέρωση οι ε, φόροι μειώνονται με αποτέλεσμα να υπάρχουν ε, μειωμένα ε, κρατικά έσοδα και κατά συνέπεια το κράτος δεν μπορεί να παρέχει πολιτικές υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών. Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα εντάχει να αναφέρω τις άλλες προτάσεις που κάνουμε από την ε, κοινή μας, εργασίας, ε, ε, κοινή μας εργασία. Εκτός από τα κεφάλαια ισότητας των φύλων και βιωσιμότητας θεωρούμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στις εταιρείε και θα πρέπει να περιορίσουμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα, τα την πνευματική, ε, τα πνευματικά δικαιώματα. Ε, όλα αυτά συζητώνται αυτή τη στιγμή στο ε, πλαίσιο του ΟΗΕ. Οι γυναίκες ευθύνονται ιδιαιτέρως για τα ζητήματα τροφίμων και επηρεάζονται λοιπόν από τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε, λέει η Πρόεδρος. Έχω να προσθέσω μόλις δύο προτάσεις, λέει η ομιλήτρια. Κλείνοντας λοιπόν, Πιστεύω ότι ε, τα υπόλοιπα ζητήματα έχουν αναφερθεί ήδη από τις προηγούμενες ομιλητρίες, οπότε θα ολοκληρώσω εδώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μάγερς ε, και τώρα ε, χαίρομαι ε, ιδιαίτερος που μπορώ να σας παρουσιάσω την κυρία Πάολα Σουμπάκη, η οποία είναι Διευθύντρια Οικονομικής Έρευνας στο Chatham House ε, το οποίο είναι ένα από τα βασικότερα Ινστιτούτα του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις. Ε, είναι ε, ειδική σχετικά με ζητήματα διεθνούς νομισματικής και σήμερα θα μας παρουσιάσει σχετικά με το πώς η πολιτική δημοσιών συμβάσεων μπορεί να συμπεριλάβει περισσότερο το ζήτημα φίλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου. Θα ασχοληθώ κυρίως με τις δημόσιες προμήθειες και τι ρόλο μπορούν να παίξουν στην κοινωνική πολιτική. Είναι πολύ ισχυρό εργαλείο. Εντάξει, μπορεί να είναι τεχνικό το θέμα, δεν είναι πολύ ελκυστικό, αλλά παρόλα αυτά. Όλη αυτή η εργασία έχει γίνει στα πλαίσια της ομάδας ε, γυναίκες για το 2020, το οποίο θέλει να βοηθήσει τις γυναίκες να μετάσχουν ε, περισσότερο στην οικονομική ζωή, ούτω ώστε να υπάρξει μια ανάπτυξη ισότιμη για όλους. Ε, οι δημόσιες ε, προμήθειες εκτιμώνται από την Διεθνή Τράπεζα στα 13 εκατομμύρια. Είναι γύρω στο 30% στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ στις αναπτυγμένες γύρω στο 10%. Παρ' όλα αυτά, ενώ είναι τόσο μεγάλη αυτή η αγορά, μόνο 1% παρέχεται από γυναίκες, από, επιχειρημα... από επιχειρηματίες που είναι γυναίκες. Και θα αναφερθώ σε αυτό που είπαν και οι προηγούμενες. Τι σημασία παίζουν οι δημόσιες προμήθειες, τι ρόλο παίζουν για την πρόθεση της ε, ισότητας των φύλων. Ιδιαίτερα η συμμετοχή στις δημόσιες προμήθειες μιας χώρας θα πρέπει να είναι η δυνατότητα για να συμμετάσχουν οι γυναίκες ε, στο εμπόριο και τις εξαγωγές. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με αυτό. Για παράδειγμα, πολύ συχνά είναι πολύ περίπλοκες οι διαδικασίες ε, για να συμμετάσχει κανείς ε, σε μια διαδικασία για μια σύμβαση για παροχή δημοσίων προμηθειών. Οπότε δεν είναι εύκολο να συμμετάσχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως ε, δραστηριοποιούνται οι γυναίκες επιχειρηματίες. Μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε μέτρα για να γίνουν αλλαγές. Ιδιαίτερα προτείνουμε σε μια έκθεση που θα δημοσιεύσουμε σε κάποιες εβδομάδες, προτείνουμε μία προσέγγιση που περιέχει τρία σημεία. Και οι κυβερνήσεις αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί που συνάπτουν συμβάσεις μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα μέτρα. Πρώτο λοιπόν, πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δημόσιες προμήθειες για να βοηθήσουμε τις γυναίκες να ξεπεράσουν τα εμπόδια για να συμμετάσχουν στην οικονομία. Ξεκινάμε λοιπόν σε αυτή την έκθεση εξετάζοντας γιατί σε κάποιους τομείς κατασκευές, δημόσια έργα, εξόριξη, χρηματοπιστωτικός τομέας όπου δεν ε, υπάρχουν πολλές γυναίκες. Είναι από την πλευρά της προσφοράς ή της ζήτησης. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν ούτως ώστε περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν σε αυτούς τους τομείς να αυξηθεί έστω και λίγο ο αριθμός των γυναικών που ασχολούνται σε αυτούς τους τομείς. Το δεύτερο στοιχείο της δέσμης μας είναι να καταργήσουμε τους φραγμούς για τις δημόσιες προμήθειες, για τις επιχειρήσεις, των οποίων ηγούνται οι γυναίκες. Και τρίτον, να αυξηθεί η διαφάνεια όλης της διαδικασίας. Προτείνουμε, για παράδειγμα, ότι οι επιχειρήσεις που κάνουν προσφορές για δημόσιες συμβάσεις και είναι μια σύσταση που μπορεί να μπει και σε εμπορικές συμφωνίες αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφίστανται έλεγχο για το κατά πόσον εκπροσωπούνται διάφορες ομάδες του πληθυσμού στο εργατικό του δυναμικό αν ε, υπάρχουν καλές πρακτικές για ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών και θα πρέπει να είναι και διαφανείς να δίνουν στοιχεία για το αν υπάρχουν διαφορές στις αμοιβέ ε, των ανδρών ε, σε σχέση με τις αμοιβέ των γυναικών στο προσωπικό τους. Οι δημόσιες προμήθειες λοιπόν είναι ένα μέσο για να επιταχύνουμε αλλαγές. Έτσι θεωρούμε. Τώρα, μελετήσαμε ορισμένες περιπτώσεις χωρών που εφήρμοσαν ορισμένες από αυτές τις πολιτικές που μπορούν να μας βοηθήσουν να εξαγάγουμε διδάγματα για θέματα εμπορικών συμφωνιών, όπως είπαν και οι προηγούμενες. Ορισμένες χώρες όπως η Νότια Αφρική και η Αυστραλία έχουν, έχουν αξιοποιήσει τις δημόσιες προμήθειες για να ε, βοηθήσουν ε, κάποια τμήματα του πληθυσμού, κάποιες κοινότητες Μπορούν λοιπόν να αξιοποιηθούν για να βοηθήσουν και τις γυναίκες να συμμετάσχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. Στη Χιλή για παράδειγμα. Υπάρχει πρωτοβουλία Chile Compra, δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, τις οποίες διοικούν γυναίκες στηρίζονται και βοηθούνται και τους παρέχεται κατάρτιση για να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, για δημόσιες προμήθειες. Επίσης, οι πολιτικές αυτές δεν ε, σημαίνει ότι πρέπει ε, να ευνοούν τις γυναίκες. Όχι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που θα βοηθάει, θα στηρίζει, θα καταρτίζει τις γυναίκες για να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά βέβαια εντάξει, υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα. Ίσως στην ε, αρχή θα πρέπει να τις προωθήσουμε, να τις ευνοήσουμε ως ένα πρώτο βήμα. Αλλά από πλευράς αρχής απλώς τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, να ανταγωνιστούν τις άλλες εταιρείε. Δεν θέλουμε να υπάρχει ένας ειδικό τομέα για τον οποίο να επιτρέπεται ας πούμε να συμμετάσχουν μόνο γυναίκες στην υποβολή προσφορών. Σημασία έχει επίσης η έρευνα και κοινή μεθοδολογία για τη συλλογή στοιχείων. Τα στοιχεία είναι πολύ κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε ποιες εταιρείε συμμετάσχουν, σε ποιες διαδικασίες προσφορών. Θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργούν αυτές οι αγορές των δημοσίων προμηθειών. Επίσης πρέπει να έχουμε και σαφείς ορισμούς. Τι σημαίνει επιχείρηση που διοικείται από γυναίκα. Υπάρχει κάποιο όριο αριθμού γυναικών που συμμετέχουν σε κάποια όργανα αυτής της εταιρεία. Ιδιαίτερα για εμπορικές συμφωνίες. Πρέπει να έχουμε εναρμονισμένους ορισμούς, γιατί πρέπει να έχουμε κοινέ προδιαγραφές. Άρα πρέπει να τις ορίσουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα. Και τώρα μερικές συστάσεις. που θα περιληφθούν και στην έκθεσή μας. Οι δημόσιες προμήθειες είναι μια δυνατότητα για να συμμετάσχουν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας, αλλά και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Να συμμετάσχουν περισσότερο σε αυτή την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής αξίας, γιατί ορισμένες φορές μπορεί να ε, θίξει τα δικαιώματά τους. Δεν θα πρέπει να είναι έτσι, αλλά πρέπει να εργαστούμε για να το αποφύγουμε. Πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο οι γυναίκε επιχειρηματίε στι δημόσιες προμήθειες και πρέπει να θέσουμε σωστούς ορισμούς, πρέπει να υπάρχουν στόχοι για το πόσο θα συμμετέχουν οι γυναίκες, πρέπει επίσης να έχουμε και κάποια μητρώα για τις γυναίκες που συμμετέχουν στις δημόσιες προμήθειες, πρέπει να επεκταθεί αυτή η δυνατότητα και να απλουστευτεί και η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ορισμένα είναι, ε, ορισμένες, για παράδειγμα, διατάξεις για την υποβολή προσφορών είναι εντελώς απαράδεκτες και άχρηστες. Μπορούν να, ε, λοιπόν να καταργηθούν. Και καταλήγω. Στις εμπορικές συμφωνίες πρέπει να υπάρχουν συστάσεις για προγράμματα επενδύσεων και βοήθειας που οπωσδήποτε να ε, συμμετέχουν επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από πλευράς ε, ε, πολυπικιλότητας του προσωπικού τους και λαμβάνοντας υπόψη το, και λαμβάνουν υπόψη την ισότητα γυναικών. ο επόμενος ομιλητής μας, το ΜΑΜΠΑΡΤ, που είναι επικεφαλής της μονάδας για το εμπόριο στην Γενική Διεύθυνση Έχουμε ζητήσει να συμπεριλαμβάνονται αυτά τα θέματα στι εμπορικέ συμφωνίε τη Ένωση και την εμπορική πολιτική. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε πληροφορίε για τι ε, μεθόδου που έχει αναπτύξει η υπηρεσία του και να μα δώσετε και ορισμένα στοιχεία για τη συμφωνία με τη Χιλή για το πώ θα συμπεριληφθεί το θέμα του φίλου διαπραγματεύσει και σα παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Συμπρόεδρε. Πολλά θέματα εδώ και θέλω Επανέτα σε όλα αυτά τα σημεία που έχετε δείξει. Εμείς ήρθαμε εδώ ακριβώ ε, την προσπάθειά μας για να ληφθεί υπόψη η ισότητα των φίλων και έχω και τους συναρμόδιους συναδέλφους. Είναι σημαντικό το ζήτημα και το λαμβάνει υπόψη η Γενική Διεύθυνση για το εμπόριο. Και ξεκινώντας θα πρέπει να σας πω ότι και εμείς προσεκτικά λαμβάνει υπόψη τη λέτε και χαίρομαι που συμμετέχω εδώ σε αυτό το πάνελ με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους σας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η προβληματική και τονίζω ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για το θέμα αυτό και μπορούν να γίνουν περισσότερα από κοινού με το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου. Η κυρία Μάρστον πρόκειται να φιλοξένησε στις 20 εκτού το Διεθνές Φόρουμ για το εμπόριο και τις γυναίκες. Έτσι καταλαβαίνετε πώς ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα. Πώς θα προωθήσουμε δηλαδή την ε, υπόθεση της ισότητα και σε σχέση με την εμπορική πολιτική. Οπότε έχουμε το σχετικό θεματολόγιο για όλες μας τις πολιτικές. Όπως το ε, ζήτησαν όλοι οι εξέχοντες ε, προσκεκλημένοι μας και εσεί. Οπότε όλοι είστε προσκεκλημένοι στις 20 Ιουνίου σε αυτό το Διεθνές Φόρουμ. Η εμπορική πολιτική ε, πρέπει να διακρίνεται από ανοιχτό πνεύμα ε, και να είναι ανοιχτή και προς την τεχνολογία, προς τον κόσμο, προς ε, το κεφάλαιο και βέβαια δεν θα πρέπει να γίνονται δυσμενείς διακρίσεις σχέση με την πολιτική αυτή οπότε απριόρι μπορεί η εμπορική πολιτική να βοηθήσει την ισότητα των φίλων. Επίσης, όπως είπαν και οι ομιλητές, το να μην υπάρχει θεσμής διάκριση δεν είναι όλο το θέμα, δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Άρα αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι το τι μπορεί να κάνει η εμπορική πολιτική και οι εμπορικέ συμφωνίε για την υπόθεση τη ισότητα. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μπορεί να κάνει παραπάνω πρώτα-πρώτα. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο προαναφέρθηκε ότι θα πρέπει να το επισημάνουμε, να έχουμε δηλαδή μια εμπορική στρατηγική που να ε, διέπεται από την αρχή εμπόριο για όλους και έτσι να ωφελείται από την πολιτική μας ε, ο, ο καθένας και οι γυναίκες, όλοι όσοι εμπλέκονται. Και εχθές ε, εγκρίναμε ένα έγγραφο προβληματισμό όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης και αφορά την, το πώς θα τι θα σέψουμε την ε, παγκοσμιοποίηση, οπότε στα πλαίσια αυτά δεν θα πρέπει να φυγεί κανείς και από τους κανόνες που διέπουν το εμπόριο. Αυτό θέλουμε να εξετάσουμε πιο προσεκτικά γιατί είναι πολύ σημαντικό και από την πλευρά του να ε, τηρούμε τις βασικές αξίες μας σε σχέση με τους αναπτυσιακούς στόχους και να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρξει απασχόληση που όλα αυτά θα πρέπει να διέπουν την παγκόσμια οικονομία. Οπότε αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα και είπαμε με βάση την αρχή trade for all για την ισότητα, για τα δικαιώματα των γυναικών. Οπότε όλα αυτά βαθμία καλύφθηκαν από την αξιολόγηση της ε, εμπορικής πολιτικής μας όπως ε, το τόνισαν η μιλητέ και η κυρία Σουμπάκη. Οπότε θα πρέπει πρώτα πρώτα να καταλάβουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις από τα όσα κάνουμε και μετά να δούμε που η υπόθεση επιδέχεται βελτιώσεις. Ε, Γι' αυτό ο έρευνα της κυρίας Φοντάνα για το θέμα μας, γιατί είναι με τις ε, πρόσφατες μεγάλες εμπορικές συμφωνίες όπως η ΣΥΤΑ και άλλες, ε, που ήδη έχουν συναυθεί ή είναι τώρα υπό διαπραγμάτευση και σας τονίζω ότι πολλά από όσα κάνουμε για την αξιολόγηση της πολιτικής μας παίρνει χρόνο. Οπότε η μελέτη ήδη έχει αρχίσει για το ΣΥΤΑ αλλά και το 2011 ξεκίνησε αυτή η μελέτη για την ΣΥΤΑ αλλά έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει. Άρα αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίση έχουμε συμφωνήσει με Μαρόκο, Αρμενία για την Ισία το 2013. Η Ορδανία κλπ. Οι σχετικέ μελέτες αναγνώρισαν τις επιπτώσει τη ε, γυναίκης. Οπότε αυτές οι μελέτες επιπτώσεων θα ολοκληρωθούν φέτος όσον αφορά τα περιβαλλοντικά αγαθά να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιε είναι οι ευκαιρίε τη εμπεσόμενε χώρα για τι ε, γυναίκε, σαν απόρρια τη απορρίθμιση και απελευθέρωση. Επίση, έχουμε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Ιαπωνία και εκεί υπάρχει μια μελέτη για, για τι επιπτώσει όσον αφορά τις, τις ανισότητες και με τη Μιανμάρ έχουμε άλλη μια μελέτη για τους κινδύνους, για τις ευκαιρίες για τις γυναίκες, τι γίνεται με τις επενδύσεις για εταιρείε, οπότε Βλέπετε, σε όλη τη διαδρομή της διαδικασίας εξετάζουμε το ποιες είναι οι επιπτώσεις του τι κάνουμε και τι διαπαιδευόμαστε για τις γυναίκες. Και υπάρχει ένα σχετικό εγχειρίδιο για αυτές τις μελέτες επιπτώσεων, οπότε μπορείτε βρείτε εκεί πολλά στοιχεία. Και ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπε η κυρία Σουμπάκη για την κοινή μεθοδολογία για την έρευνα, γιατί χωρίς να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες έχουμε πολλές προκλήσεις όσον αφορά τα οικονομικά πρότυπα. Γιατί αν σε ένα οικονομικό μοντέλο έχουμε μεταβλητές που δεν ισχύουν, τότε το αποτέλεσμα θα είναι αποτυχημένο. Επομένως θα πρέπει να είναι αξιόλογα τα δεδομένα. Να, μια πρόκληση του πώς κανείς θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα πώς αυτά θα τα αναλύσουν, θα τα κατατάξουν. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά την αξιολόγηση της εμπορική πολιτικής, για να μην επαναλάβω αυτά τα οποία προείπατε, να σας πω ότι από δική μας πλευράς πολλά έχουν ήδη καλυφθεί από τις εμπορικές συμφωνίες και τα του ILO και την υλοποίησή τους του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, επίσης το πρόγραμμα GSP Plus και εκεί καλύπτεται η ισότητα, οι χώρες θα πρέπει να κυρώσουν αυτές τις συμφωνίες και έχουμε 27 ε, βασικές συνθήκες που πρέπει να κυρωθούν από όλες τις χώρες όπως επίσης και τη συμφωνία με τον Καναδά. Τώρα, τι γίνεται στα πλαίσια του ΟΣΑ όσον αφορά την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα έχουμε τη στρατηγική Aid for Trade τη βοήθεια μέσω του εμπορίου δηλαδή Θεωρούμε ότι και εδώ δίνονται ευκαιρίες όσον αφορά να καλυφθεί η υπόθεση της ισότητας των φύλων. Και έχουμε και άλλα μέσα εμπορικής πολιτικής που και αυτά βοηθάνε στην οικονομική χειραφέτηση της γυναίκας. Και τα σχετικά με τις ΜΜΕ, ξέρω ότι υπάρχουν επικρίσεις, αλλά έχουμε επίσης ότι το ITC λέει το 40% των ΜΜΕ παγκοσμίω ε, ανήκουν σε γυναίκες. Οπότε με τις εμπορικές συμφωνίες φροντίζοντας τις ε, ΜΜΕ και τις ιδιοτυπίες τους βοηθούμε και τις γυναίκες. Και πολλές φορές υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ σε συμφωνίες εμπορικές. Κάτι άλλο που δεν αναφέρθηκε είναι το τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν έχουμε εδώ για την γυναικεία χειραφέτηση ειδικέ διατάξεις, όμως συνεχώς προσπαθούμε και σε αυτό το πλαίσιο και διμερός και πολυμερός. Οπότε βοηθούμε έμεσα. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ψηφιοποίηση, την ψηφιακή τεχνολογία τέλο πάντων, ποιε είναι οι επιπτώσει στην αγορά τη απασχόληση, πώ ε, δίνονται ευκαιρίε, και πώς θα έχουμε πιο ευέλικτη απασχόληση. Πώς θα έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, πώς θα βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Να δούμε τι θα γίνει με αυτούς που δουλεύουν από το σπίτι, τι γίνεται με τις γονικές άδειε. Οπότε και εδώ μπαίνει θέμα γενικές χειραφέτησης. Τώρα, τον υπόλοιπο χρόνο. Για να δούμε κάποιες ερωτήσεις που έχουν τεθεί, τι μπορούμε να κάνουμε και τι γίνεται και με τη συμφωνία με τη Χιλή. Βέβαια δεν μπορούμε να προδικάσουμε στο τι θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Χιλή. Κύριε Μάλστρομ ήδη έχει πει και επιβεβαιώνω ότι όντω πέραν των επιπτώσεων για την ισότητα των φύλων επίσης διερευνάται το πώ μπορούμε να έχουμε κάποιε ειδικέ διατάξει για την ισότητα των φύλων. Οπότε βήμα-βήμα βελτιωνόμαστε. Άλλο σημαντικό βήμα έτσι το το πω σαν διαφήμιση είπαμε για την εκδήλωση που θα έχουμε στις 20 Ιουνίου. Αυτό θα βοηθήσει και να διαμορφωθεί η εμπορική μας πολιτική, και επίσης θα σας παρουσιάσουμε και μια σχετική έκθεση στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Το δικό μου τμήμα ασχολείται με την ε, στρατηγική Aid for Trade που θα που για αυτή τη διέτεια και όλα αυτά καλύπτουν πολλά από όσα σήμερα συζητήσαμε και θα λάβουμε υπόψη και τις απόψεις που ακούστηκαν και εν ώψη του φόρμου λοιπόν της 20 Ιουνίου Ευχαριστώ. Ε, Εμεί ευχαριστούμε όλους τους ομιλητέ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα παρατηρήσεις και ερωτήσεις από τους ε, βουλευτές. Α, θα πρέπει να αρχίσουμε από τις συνεισηγήτριε. Ευχαριστώ πολύ ειδικά τους ε, ομιλητές μας και τους καλεσμένους μας, ε, διότι ε, επεξεργασόμενοι το συγκεκριμένο θέμα κατανοούμε το πόσο σημαντικό είναι ο συγκεκριμένο τομέας και επικεντρωθήκαμε ιδιαιτέρως μέσω της ακαδημαϊκής έρευνας σε αυτό, αλλά και στα όσα έχει κάνει η κοινωνία των πολιτών. Όμως φαίνεται ότι και εσείς στην Κομισιόν έχετε φτάσει σε αυτό το θέμα, όμως και πάρα πολύ καιρό δεν αποτελούσε ζήτημα. Εμείς στο Κοινοβούλιο λοιπόν το προωθούμε προωθούμε αυτό. Ε, εργαζόμαστε ε, πάνω στην παγκόσμια λυσίδα αξίας ε, και θα λάβουμε υπόψη μας πολλά από τα όσα έχετε αναφέρει. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο στόχος μας είναι ε, να μην επικεντρωθούμε μονάχα στην ανάλυση και τα δεδομένα. Ναι, χρειάζονται όλα αυτά, όμως θα πρέπει να πάμε ακόμα πιο ε, πέρα στην έκθεσή μας και να κάνουμε πιο ε, συγκεκριμένες προτάσεις. Έχω παρατηρήσει ότι κανένας από την δεξιά και από τους φιλελεύθερους δεν είναι εδώ, διότι πολλοί εξ αυτών καθορίζουν μέσω της, των ιδεών τους την ευρωπαϊκή πολιτική, πολιτική εμπορίου και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα πρόβλημα και μία πρόκληση και θα συζητήσω με τους συναδέλφους μου. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως, αποτελεί πρόκληση. Ε, δεν έχουμε προσκληθεί ε, ε, στην, εκδήλωση της 20ης Ιουνίου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχει διορθωθεί όμως είναι ένα πρόβλημα. Ελπίζω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη εκθεσή θα μπορέσει να εξετάσει το βορρά και νότο όπως είπε η κυρία Williams τις σχέσεις βορρά και TTIP αλλά και πολυμερή την πολυμερή συμφωνία όπως είναι το ΤΙΣΑ. Έχουμε αρκετά δεδομένα εδώ πέρα ε, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, ε, τις γυναίκες ως οικονομικοί παράγοντες και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και στο ε, ζήτημα των νομοθετών και το, την ικανότητα που έχουν στο μέλλον να ρυθμίζουν. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, χτίσουμε πάνω σε όλο αυτό σχετικά με το ότι οτιδήποτε είναι ανοιχτό, είναι καλό. Το είχαμε αυτό όμως, την αλλάξαμε διότι δεν συμφωνούσαμε τα δεδομένα που είχαμε. Πολλά θα πρέπει να αλλάξουν στην εμπορική πολιτική. Αυτή είναι η υπεποίθησή μου και θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου εδώ αλλά και στην Επιτροπή Ίντα. Έχουμε αλλάξει πολιτικής δημοσίων συμφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και το πώς Εξετάζουμε τις αρχές των μη διακρίσεων, ούτω ώστε να επικεντρωθούμε στην ισότητα των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη. Θα ήθελα επίσης να ακούσω από εσά σχετικά με αυτό το εργαλείο το οποίο συζητά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ε, αξιολόγηση επιπτώσεων πάνω στην ε, βιωσιμότητα ε, και επιπρόσθετα κάποιοι από εσάς αναφέρατε ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, τομέων να προστατεύονται ή να υπάρχει μια καθυστέρηση ε, ώστε να απελευθερώνονται. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποιους τομείς έχετε υπόψη σας και θα επανέλθω σε εσάς καθώς καταρτίζουμε την έκθεσή, σας, την έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ πριν επιστρέψουμε στους ε, ομιλητές θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Φορέντσα. Ευχαριστώ και εγώ τους εξέχοντες προσκεκλημένους μας. Θα βοηθούμε πολύ στο έργο μας από τα όσα μας είπανε και εγώ και η Björk. Αυτά τα σχετικά επομένως για το Διεθνή Συμπόριο, αλλά επίσης ε, ε, εκτός από την αρμόδια επιτροπή, ε, και η δική μας επιτροπή των γυναικών. Ασχολούμαστε με το mainstream, οπότε αυτή η προσπάθεια της η δική μου, της κυρίας Björk, ε, θεωρούμε ότι μπορούμε και οφείλουμε να συνεργαστούμε οι δύο επιτροπές από κοινού ε, και όλο ένα περισσότερο να συνεργαζόμαστε γιατί νομίζω ότι φάνηκε σήμερα από τα όσα ακούσαμε για πολλωστή φορά αυτό που θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδους προοπτική ουδέτερη όσον αφορά τα δύο φύλλα και να μην είναι τυφλή η πολιτική όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Και ακόμα καλύτερα να υπάρχει ευαισθησία στην υπόθεση της ισότητας των ε, φύλων και στην εμπορική πολιτική. Θέλω να σας προσθέσω τώρα τα εξή. Είναι σημαντικό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει υλοποίηση σε αυτές τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Και συμφωνώ με αυτά που είπε η Μπιόρκ. γιατί στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής εξεπλάγει όταν είδα ότι δεν είχε ληφθεί υπόψη ο δικός μας ρόλος των δύο συνεισηγητριών. Οπότε από αυτής της πλευράς είναι σωστό να υπάρξει κάποιο είδου αποκατάσταση της κατάστασης και από το gender blind να πάμε στο gender sensitive. Να υπάρχει δηλαδή ευαισθησία στο πρόβλημα της ισότητας. Να υπάρξει βούληση. Να ληφθεί η υπόθεσή μας στην εμπορική πολιτική αλλά και στην εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση της πολιτικής αυτής επίσης και όσον αφορά το πώς θα περιχαρκώσουμε ένα άλλο θέμα. Κάτι το οποίο θίγω στο κείμενό μου. Για τη σχέση μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπορικής πολιτικής. Δηλαδή, αφενό θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη τα γυναικεία δικαιώματα, όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και πάντοτε θα πρέπει οι σχετικέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να λαμβάνονται υπόψη και να περιέχονται ει τι εμπορικέ συμφωνίε. Βλέπουμε τώρα συμφωνίε, βλέπουμε μια πολιτική που θα πρέπει να θεωρεί δεσμευτικά τα των επενδυτών. Και επίσης να είναι δεσμευτικά όλα όσο έχουν σχέση με την στην πράξη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Α, να σα προσθέσω και κάτι άλλο. Ακούσαμε πολλά για το πώς θα πρέπει να την υπόψη η ισότητα των φύλων παντού και αυτό αφορά όλους τους τομείς. να καλυφθούν υπόψη οι μετανάστες, οι γυναίκες, οι άντρες, οι ΛΟΑΔ. Και έτσι να ληφθεί υπόψη και η πολιτική διάσταση. Φεμινιστικό κίνημα, ούτω ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την αδιαφορία προς την υποθεσιότητα στο φίλο των gender blind. Τώρα, εν κατακλείδη, να σας πω για τις ανισότητες. Πολλές φορές όταν ε, ορίζουμε τις οικονομικές παραμέτρους δεν λαμβάνει υπόψη τις ανισότητες. Ξέρουμε ότι ε, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αυτό το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών. Πάμε περίπου στο 16% του πραγματικού μισθού και φτάνει στο 40% όσον αφορά το εισόδημα σε διάφορους ε, τομείς ε, όπως σε αυτές τις υπηρεσίες φροντίδας όπου δεν ασχολούνται πολλοί άντρες και πολλές φορές σε αυτούς τους τομείς όμως η ανεργία περισσότερο θίγει τις γυναίκες και άρα έχουμε κάποια μέτρα που θίγουν τις γυναίκες σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν σχετικέ συλλογικέ ρυθμίσει. Και πάλι όμως να ευχαριστήσω για όλες τις εισηγήσει που ακούσαμε. Και θέλω να σας πω για τις απαντήσεις που θα δώσετε ότι συμφωνούμε στα περισσότερα σημεία να, όσον αφορά δηλαδή με ποια μέσα θεωρείτε να μας πείτε ότι μπορούν να βοηθήσουν εάν τα εντάξουμε στο κείμενο του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. Εμείς δηλαδή έτσι να βάλουμε το λιθαράκι μας. Οπότε να μας πείτε το τι πρέπει να προτάξουμε θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Και πάλι σας ευχαριστώ για τις αναλύσεις σας. Um, Ευχαριστώ πολύ ε, τις συνεχιστηγήτριες. Τελειώνει ο χρόνος μας όμως και ξέρω ότι όλοι θέλουν κάτι να προσθέσουν. Γι' αυτό το λόγο, ε, μπορεί, αν μπορείτε να περιοριστείτε στο ένα λεπτό, ε, διότι θα πρέπει να έχουμε τελειώσει στις 11.30. Ε, αρχικά θα δώσω το λόγο στην Χάιντι και ε, στη συνέχεια θα περάσουμε προς όλους τους κοιόδες που βρίσκονται εδώ. Ευχαριστώ. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη όπως ε, ζήτησες, λέει στην πρόεδρο. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε το ε, κατά πόσο το εμπόριο έχει ε, μια διάσταση φύλου και κατά πόσο θα πρέπει να προωθήσουμε την εφαρμογή αυτού. Θα πρότεινα στην, στο Digitrade Trade να παράσχει εκπαίδευση πάνω σε αυτά τα ζητήματα και όχι μονάχα να περιοριστεί στις υπηρεσίε που ασχολούνται με, την, με το mainstream του φύλου θα ήθελα να επικεντρώσω το ερώτημά μου στο ζήτημα του νότου ε, όσον αφορά ε, τα σχόλια της ε, κυρίας Williams για τις εμπορικές συμφωνίες και το πώς αυτές επηρεάζουν τις, τις τοπικές κοινωνίες ε, και πώς μπορούμε να εξετάσουμε την ε, επιρροή του φύλου πάνω σε αυτές τις συμφωνίες οι οποίες δέχονται τόσο μεγάλη κριτική. Ευχαριστώ ε, Χάιντι. Θα ήθελε τώρα κάποιος άλλος να κάνει κάποιο σχόλιο. Ροντρίγκες Πινιέρο, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ όλες τις ομιλήτρες και να σας συγχαρώ και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την κοινή αυτή συνεδρίασή μας, τις δύο επιτροπές που πρέπει να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε το εμπόριο πραγματικά να συμπεριλάβει προοπτική φύλου. Αναγνωρίζω ότι η Επιτροπή ε, έχει ευαισθητοποιηθεί. Όταν ήρθα τον Ιούλιο του 2014 στο Κοινοβούλιο, έλεγαν ότι οι συμφωνίες αυτές είναι ουδέτερες από πλευράς φίλου. Άλλαξε αυτό τώρα. Κατάλαβαν ότι έχει σημαντική διάσταση φίλου η εμπορική πολιτική. Τώρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσει περιεχόμενο η εμπορική πολιτική, περιεχόμενο προοπτικής φίλου. Η συζήτηση με τη Χιλή είναι μια ευκαιρία γιατί η Χιλή είναι μια χώρα που όντως ε, αποδέχεται ότι έχει διάσταση φίλου το εμπόριο. Αλλά δεν πρέπει απλώς να την αναφέρουμε την προοπτική φύλου. Πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο περιεχόμενο, ένα κεφάλαιο για την διάσταση φύλου και να συμμετάσχουμε οι εμπειρογνώμονες και το Κοινοβούλιο ούτως ώστε να έχει την μέγιστη, ε, το μέγιστο περιεχόμενο και κυρίως τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Μια πρόταση. Εάν δεν έχετε εμπειρογνώμονες φύλου στη διαδικασία διαπραγματεύσεων από την αρχή για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική διάσταση στις ε, συζητήσεις. Γιατί ναι, μεν πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο φίλου, αλλά είναι το θέμα κάτι που αφορά όλους τους τομείς μια εμπορική συμφωνίας. Πρέπει όντως, ε, μόνο έτσι μπορούμε να αποφύγουμε αρνητικέ επιπτώσει και έτσι θα αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό των γυναικών. Να έχετε λοιπόν μαζί σας σε όλη τη φάση της διαπραγμάτευσης ειδικού για τα θέματα φύλου και μετά και στις μελέτες αντικτύπου και εξ άντε και εξ post. Γιατί εάν, ε, όπως είπε μία από τις ομιλήτρες, αν δεν έχετε ένα κατάλογο των ευαίσθητων ε, τομέων για κάθε χώρα, για κάθε συμφωνία, όπου είναι πιο ευαίσθητες οι γυναίκες και όπου πρέπει να γίνουν περισσότερα για να τις βοηθήσουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το εξάντε. Αλλά κατόπιν πρέπει να έχουμε μια καλή παρακολούθηση και αξιολόγηση. Εξορισμών δεν ωφελεί. Γιατί δεν θα διορθώσουμε τα λάθη. Δεν θα ε, προωθήσουμε το δυναμικό των γυναικών. Γι' αυτό κάνω έκκληση από την αρχή να τα λαμβάνετε υπόψη. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τις γυναίκες. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ε, για, πολύ σύντομα παρακαλώ. Η Μαρία. Έχω κάποιες ερωτήσεις και στην Επιτροπή και στις διάφορες ομιλήτριες. Η πρώτη ερώτηση προς την Επιτροπή. Οι συνθήκες αυτές, οι συνθήκες οι ευρωπαϊκές επιβάλλουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εμπορική της πολιτική. Πώς σέβεται η Επιτροπή. Τι μέσα έχει η Επιτροπή για να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν υπάρχουν κατάφορες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών σε κάποιες χώρες. Είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει μέτρα για να το διορθώσουν. Και ποια. η μελέτε που το είδαμε εδώ στην Επιτροπή Γυναικών. Είχαμε μια μελέτη που μας έλεγε ότι στις μελέτες αντικτύπου τη Κομισιόν δεν υπήρχε καμία γυναίκα ερευνήτρια. Άλλαξε αυτή η κατάσταση υπάρχουν και γυναίκες ερευνήτριες που να συμμετέχουν στις μελέτες αντικτύπου και τι κάνετε για να τις ε, ευνοήσετε. Γιατί πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία, ίσως ποσοστώσεις, για να υπάρχουν οπωσδήποτε γυναίκες, περισσότερες. Επίσης, οι μελέτες αντικτύπου έχουν και μηχανισμούς παρακολούθησης μετά. Πώς λειτουργούν αυτές ε, οι διαδικασίες, γιατί δεν ξέρουμε. Όπω είπε και η Όλυν προηγουμένως, αφορά και τις σχέσεις νότου-νότου. Ε, συγγνώμη, βορρά-βορρά. Αλλά όχι μόνο. Βορρά-βορρά, για παράδειγμα. Η ΣΕΤΑ. Σήμερα στην Ευρώπη συζητάμε για την ισορροπία επαγγελματική και ιδιωτική ζωής. Πώς δηλαδή να υπάρχει επαρκής κοινωνική προστασία για να επιτρέπουμε στις οικογένειε να λειτουργούν. πώ μια εμπορική συμφωνία με έναν εταίρο όπω ο Καναδά, που είναι φιλική χώρα που έχει κοινωνικές ε, παροχές ε, ισότιμες περίπου. Πώς πρέπει να αποφύγουμε το να λέμε μειώνεται η ανταγωνιστικότητά μας ε, επειδή δίνουμε προστασία στις οικογένειες. Υπάρχει στον Καναδά για παράδειγμα μία διαδικασία, υπάρχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει να υπάρχει κινητικότητα των γυναικών. Άρα Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απόσπαση γυναικών από τον Καναδά που να έρχονται να εργάζονται εδώ. Και αυτό σημαίνει μετά ότι θα υποστούμε πίεση από τις ε, οργανώσεις των γυναικών και εμείς φυσικά ε, θέλουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Πώς είναι δυνατό σε μια εμπορική συμφωνία να αποφύγουμε αυτό το, το κοινωνικό ντάμπινγκ και για τις σχέσεις Προφανώς είναι σημαντική η διάσταση των γυναικών. Στις διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών με την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Ασία, οι κύριοι εταίροι και συνομιλητέ μας είναι οι εξαγωγικές βιομηχανίες. Όταν συζητάτε με την Κάνα, τότε κυρίως ο τομέας της μπανάνας ε, είναι ο συνομιλητής μας. Οι γυναίκες που εργάζονται στην ε, τοπική γεωργία για την παραγωγή τροφίμων που καταναλώνται τοπικά δεν συμμετέχουν. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις που εξάγουν μπανάνες, που φυσικά δεν θέλουμε να τις στήξουμε, είναι οι βιομηχανίε, που καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα τη καλλιεργής γη και δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να έχουν γεωργία μικρής κλίμακας. Δεν συμμετέχουν οι γυναίκες. Πήγαμε, συναντηθήκαμε στους οργανώσεις γυναικών εκεί, ποτέ δεν τις ρωτήσανε για τη γνώμη του για τι εμπορικέ συμφωνίες με την Κάνα. Ούτε οι γυναίκες που εργάζονται και επιτόπου, ούτε οι γυναίκε βουλευτέ που εργάζονται για τα δικαιώματα των γυναικών έχουν καμία συμβολή. Αυτό αφορά την Κάνα, το Μερκοσούρ, όλε τι εμπορικέ συμφωνίε. Δεν τι ρωτάνε. Ενώ είναι τα πρώτα θύματα αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Πώ μπορούμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Και τρίτον, έχουμε μια ζήτηση για τι γενικευμένε προτιμήσει συν. GSP συν. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό όργανο για να δώσει πρόσβαση βεβαίω. Στι ε, Ευρωπαϊκέ αγορές αλλά για αυτούς που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώ μπορούμε να έχουμε περισσότερες διατάξεις GSP συν γιατί συμπεριλαμβάνουν το φύλλο. Γιατί από τις 27 χώρες μέλη μόνο μία ε, αναφέρεται στο θέμα της ισότητας ε, των αμοιβών. Πρέπει να μπει το θέμα αυτό περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω όσους από τους προσκεκλημένους μας θέλουν να απαντήσουν σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, εάν ε, θα ήθελαν να το κάνουν. Έχουμε ένα πεντάλεπτο περίπου. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο για τα θέματα που τέθηκαν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Williams. Ήταν πολύ εύτοκε και βοήθησαν πολύ αυτέ οι ερωτήσεις. Έχω κάτι, ε, ε, κάτι άλλο να το δώσω στη γραμματεία να σα το μοιράσει. Τώρα για αυτό που για του τομεί που χρήζουν προστασία έχει γίνει από του ακριβιστέ πολλή δουλειά από τον ΠΟΕ δηλαδή για το πώ θα διαμορφωθεί ο τομέα των κρατικών, των κοινών υπηρεσιών όπω το νερό κλπ διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Εδώ υπάγονται κάποιες κατηγορίες που κυρίως ε, ε, αφορούν γυναίκες που εκεί δουλεύουν. Τέλο πάντων, σημαντικά θέματα και για τη διατροφική ασφάλεια. Εδώ, εδώ είναι, υπάρχουν πολλά θέματα. Νο, και σε διεθνέ επίπεδο για την παροχή υπηρεσιών θα πρέπει κάτι να γίνει. Και τώρα, όσον αφορά τι συμφωνίε οικονομικών εταιρικών σχέσεων, ΕΠΑ, ε, είπαμε ότι, ότι πιέστηκαν να τις προσφοράψουν οι Αφρικανοί. Επομένως, φέρει ευθύνη τώρα η Ευρώπη, φέρει ευθύνη η Κομισιόν. Θα πρέπει να παρακολουθήσει τις επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων και ιδίω των γυναικών και των μικροκαλλιγετών Αυτές οι συμφωνίες ΕΠΑ έχουν το δικό τους θεματολόγιο για περαιτέρω απορρίθμιση του τομέα των υπηρεσιών. Άρα αυτό παρακολουθήστε το. Να δείτε τι επιπτώσεις θα έχει. Ε, υπάρχουν ε, οι προκλήσεις οι ανεπτυξιακές και οι ρυθμίσεις σχετικές με ζωντασμούς πολλές φορές κρύβουν κινδύνους για τις ε, μικρές επιχειρήσεις. Ιδίως υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, Ανατολική Αφρική κυρίως, όσον αφορά κάποιου είδους δασμολογικέ απαλλαγέ για τις αγωγές και τώρα. Στη ΣΕΠΑ υπάρχουν κάποιες διατάξεις ευεργετικές αλλά είναι ανεπαρκείς. Υπάρχουν προβλήματα επίση με την εφαρμογή της συμφωνίας. Υπάρχουν αιρεσιμότητε, υπάρχει το θέμα του αν μπορεί να υπάρχουν άλλου είδους ε, έσοδα, ε, έχουμε κάποιους επιθετικούς ΦΠΑ, άρα θα πρέπει να επεξεργαστεί κανείς περαιτέρω αυτές τις συμφωνίες. Αυτή, αυτή τη διάσταση να την κοιτάξουμε, το τι γίνεται με τι επιπτώσει των ΕΠΑ στα δύο φύλλα. Ο Μπάρτ. Σα το λόγο. Σας ευχαριστώ για όλα όσα είπατε. Όλα, όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη, όλες σας τις προτάσεις. Δεν έχω χρόνο όμως να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά να τα πούμε. Ε, μου, κυρία Ρένα, για να φύξω ορισμένα από αυτά που αναφέρθηκαν. Κύριε Ροντρικης Πινιέρο είπε κάποια ενδιαφέροντα ότι δεν θα πρέπει να ποντάρουν Σβήνει το μικρόφωνο του ομιλητή και δεν ακούμε τι λέει. Okay. Δεν δουλεύει. Α, μάλιστα. Είπαμε ότι δεν θα πρέπει όλοι μας οι ελπίδες να στηρίζονται σε συγκεκριμένο κομμάτι συμφωνίας. Ναι, ναι, θα πρέπει να υπάρχει main statement και να εξασφαλίσουμε το ότι το θέμα της ισότητας να διαπνέει όλες τις ε, συμφωνίες, όλα τα κεφάλαια μιας συμφωνίας. Η εφαρμογή όπως αναφέρατε, ναι, το, το ξέχασα στην αρχή. Είναι πολύ σημαντικό, φυσικά. Βέβαια και μας απασχολούν στη γενική μας διεύθυνση. Η εφαρμογή των συμφωνιών είναι κάτι το πολύ σημαντικό και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε καταβάλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες για μια στρατηγική ορθής εφαρμογής. Νομίζω σας καλύπτω εδώ κυρία Άρενα για το αυτό που ρωτήσατε. Γι' αυτό έχουμε και τι επιπτώσεων. Οπότε, άπαξ και κλειστή μια συμφωνία, αρχίζει ο διάλογος με τι χώρε αντισυμβαλωμένου. Οπότε ξεκινάει μια πλατφόρμα για περαιτέρω προσπάθειε. Ε, βέβαια και δεσμευόμαστε από τη συνθήκη τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει αυτό να δει από την εξωτερική δράση, υπάρχουν πολιτικές ε, ρήτρες στις συμφωνίες και μπορεί να φτάσουμε μέχρι την αναστολή των συμπεφωνημένων εάν παραβιάζονται οι σχετικές ρήτρες. Δεν ήξερα, δεν το είχα υπόψη αυτό το οποίο είπατε εσείς για τις ερευνήτριες και τη συμμετοχή τους στις μελέτες επιπτώσεων. Ε, βέβαια όλα αυτά γίνονται από τη βάση κανόνων δεσμευτικών στη βάση προσφορών, των διαγωνισμών που κάνουμε για να προσλάβουμε. Όχι, δεν υπάρχει πάντως κάποιος κανόνας που να ευνοεί τον μεν και όχι τον δε. Είναι οι κανόνες οριζόντιοι. Μα το είπαν εδώ και οι ομιλήτρες. Ναι, φυσικά και δεν προχωρούμε σε συμβάσεις με εταιρείε που έχουν μόνο άντρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, θα το σκεφτούμε και αυτό. είναι με την κινητικότητα των εργαζομένων. Λέμε για παροχή υπηρεσιών προς τρίτες χώρες ε, και εδώ οι σχετικές συμφωνίες θα κάποιους κανόνες να λέμε τη χώρα προορισμού να βάλουμε υπόψη τον ελάχιστο μισθό να βάλουμε υπόψη το τι ισχύει γενικότερα στη χώρα προορισμού και η παροχή των υπηρεσιών πρέπει να είναι σύντονη με αυτά που σας είπα. Ευχαρίστως να τα ξανασυζητήσουμε. Αλλά θα τα πούμε και στο φόρουμ. Ήδη έχουμε κλείσει τρεις ομιλητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Και από τις δύο επιτροπές. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Θα είστε... Κυρία Φοντάνα, η τελευταία που θα το λόγο από το πάνελ. Ευχαριστώ πολύ ε, για ε, όλα αυτά τα σχόλια για αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να απαντήσω ε, σε ένα ερώτημα σχετικά με την ε, ποιότητα της ε, αξιολόγησης αντικτύπου στη βιωσιμότητα. Ναι, τα έχω διαβάσει όλα αυτά, όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την ποιότητα αυτών των αξιολογήσεων, καθώς επίσης και το εύρος, κατά το οποίο λαμβάνεται υπόψη το ζήτημα του φύλου. Ορισμένοι ε, μπορεί να το λαμβάνουν υπόψη τους, άλλοι πάλι δεν έχουν καμία αναφορά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Σε σχέση τώρα με αυτό, επίσης θα ήθελα να κάνω δύο προτάσει Αφενός, ε, είναι σημαντικό ε, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο για την ανάλυση δεδομένων. Όχι, δεν χρειαζόμαστε μονάχα ε, περισσότερα δεδομένα με βάση το φύλλο, αλλά χρειαζόμαστε και μεγαλύτερη ανάλυση. Μπορούμε να κάνουμε αρκετά με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε σε περίπτωση που υπάρχει, υπάρχει γνώση ανάλυσης δεδομένων με βάση τον, το φύλλο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν οι ικανότητες για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τα δεδομένα και αφετέρου ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σχόλιο που έγινε από αρκετούς ομιλητές ε, το οποίο είναι να αποφύγουμε την σιωπηρή προσέγγιση. Υπάρχει μία τάση να απευθυνόμαστε σε ζητήματα ε, φύλου αναλύοντας μονάχα έναν τομέα. Ο τομέας των υφασμάτων βέβαια είναι ο πιο κλασικός εξ αυτών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, το συμπεριλάβουμε γραπτό όλο αυτό και να υπάρχει μια πιο ε, συνολική προσέγγιση εξετάζοντας σε διάφορα επίπεδα το ζήτημα φύλου. Για παράδειγμα, ε, θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις ε, γυναίκες επιχειρηματίες, ε, επιχειρηματίες για δυνατότητα απασχολησιμότητας. Ταυτόχρονα όμως μειώνουμε την δυνατότητα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Τους προσφέρουμε δηλαδή από τη μία μία ευκαιρία, από την άλλη όμως τους αφαιρούμε μια άλλη δυνατότητα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε την ε, επίπτωση του εμπόριου, να έχουμε μια πιο ενιαία προσέγγιση εξετάζοντας τη διάσταση του φίλου σε όλα αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχουν τονίσει ήδη και άλλοι ομιλητές. Ευχαριστούμε. Ε, και εδώ τελειώνει η συγκεκριμένη ακρόαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που παρευρέθηκαν εδώ ε, και που ήταν τόσο συγκεκριμένοι λέγοντάς μας, ε, δίνοντάς μας πληροφορίες για τα όσα συμβαίνουν σε αυτό το τομέα. Ε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό διότι ε, δεν αφορούσε μόνο την Επιτροπή Ίντα. Όλο αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα. Ε, στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια ε, ανταλλαγή απόψεων πάνω στο έγγραφο εργασίας το οποίο θα λάβει χώρα στις 19 Ιουνίου. Εδώ λίγη συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ.